I would like to start the committee meeting, even though there are very few members in the room. Ξεκινήσουμε με τη συνεδρίαση, παρότι είναι λίγοι οι παρόντες τα μέλη. Καθίστε παρακαλώ όσοι είσαστε παρόντες. Ξεκινάμε με την ημερήσια διάταξη που σας είναι γνωστή και νομίζω εγκρίνεται ως έχει. Πρακτικά των συνεδριάσεων Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου έχουν διανεμηθεί. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρείται ότι κυρώνονται, εγκρίνονται και αυτά. Να σας ενημερώσω επίσης ότι η, έκθεση για την, η ψήφιση για την έκθεση Frontex θα γίνει την Δευτέρα 16 του μήνα από τις 6 το απόγευμα 18.00 θα είναι μακρότερη η ε, ψήφιση, η ψηφοφορία, γιατί έχουμε 195 τροπολογίες. Να σας υπενθυμίσω και για το, το κοινό σεμινάριο ε, μεταξύ της δικής μας και της άλλης κοινοβουλευτικής επιτροπής ε, που θα διεξαχθεί το Δεκέμβριο και με το πρόγραμμα το οποίο θα γνωστοποιηθεί. Άλλα διάφορα, δεν υπάρχει κανείς για τα διάφορα. Συνεχίζουμε λοιπόν ενημερωτικά η, η εξέταση στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, την προηγούμενη εβδομάδα κατά την πράσινη εβδομάδα. Πρώτον, επιτρέψτε μου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στη γραμματεία και ιδιαίτερα προς την Κλέρ που δεν παρίσταται δυστυχώς όμως πρέπει να διαβιβαστεί προς εκείνη το μήνυμα ότι ήταν εξαιρετική δουλειά που έκανε προετοιμάζοντας την αποστολή μας, την επίσκεψη αυτή που ήταν ιδιαίτερα γόνιμη συνολικά. Εγώ προέδρευα και η αναφορά σε σχέση με αυτή την έκθεση θα σας διαβιβαστεί. Είμαστε οκτώ που πήγαμε και όπως γνωρίζετε στόχος ήταν ουσιαστικά όχι να ανταλλάξουμε απόψεις με αναφερόμενους αλλά με όσους εμπλεκόντουσαν για το θέμα της ε, υιοθέτηση χωρίς ε, την γονική έγκριση στο Ηνωμένο Βασίλειο και καταχρηστική τοποθέτηση παιδιών σε ε, ανάδοχες οικογένειες, πάλι χωρίς γονεϊκή ε, άδεια και έγκριση και στην ε, Αγγλία και την Ουαλία. Πολλά παιδιά, πάνω από 5.000 πέρυσι βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση προσιοθεσία. Και αυτό μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες δύο χώρες που επιτρέπεται η μη εγκεκριμένη από τους γονείς η υιοθεσία. Θέλαμε να μάθουμε περισσότερα στοιχεία και για τους υψηλούς αυτούς αριθμούς περιπτώσεων υιοθεσιών. Ήταν σύντομη η επίσκεψή μας, είχαμε όμως την ευκαιρία να συναντήσουμε ευρύτερο φάσμα πραγματογνωμόνων και εμπλεκόμενων. Συναντήσαμε και κοινωνικούς λειτουργούς, δημοσιογράφους, εκπροσώπους συλλόγων και ενώσεων ψυχολόγων και όσους συνεπικουρούν τους γονείς. Συναντήσαμε επίσης εκπροσώπους των αστυνομικών υπηρεσιών, ακόμα και της Scotland και <clears throat> τον πρόεδρο της, ε, των θεμάτων οικογενειακής ε, δικαιοσύνης ε, που υιοθετεί απόλυτα διαφορετική θέση από τους προκατόχους του συναντήσαμε και τους ε, Βουλγάρους ε, και Λετωνούς ε, διπλωματικούς εκπροσώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξειδικευμένους δικηγόρους για τα θέματα οικογενειακού δικαίου και επίσης εκείνους που είχαν δραστήρια συμμετάσχει σε εκστρατείες για τα θέματα της οικογενειακής συνοχής και έτσι λοιπόν αντιμετωπίζαμε <clears throat> ουσιαστικά σχεδόν απόλυτα διαμετρικά αντίθετες θέσεις και απόψεις αλλά χάρη στην δυνατότητα που είχαμε μπορέσαμε να έχουμε μια σύνθετη εικόνα που αποκτήσαμε με ανταλλαγές από όλους, με όλους τους εμπλεκόμενους και θα υπάρχει δυνατότητα νομίζω να συναθούν και κάποια συμπεράσματα μετά από την εξοικείωση με το έγγραφο εργασίας που θα διαβιβαστεί. Ολοκληρώνω επαναλαμβάνοντας ότι ήταν πολύ γόνιμη και ενδιαφέρουσα η επίσκεψή μας αυτή εκεί. Μια και ήταν και η πρώτη εξεταστική τέτοια αποστολή αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας έθεσε τον πύχη υψηλά για τους όρους αποτελεσματικότητας, ποιότητας της συμμετοχής και της επιμελητίας. Η Κλέτο απαρίσταται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική δουλειά που κάνατε σε σχέση με αυτή την αποστολή και προσβλέπουμε, αδειμονούμε να δούμε το έγγραφο εργασίας όταν θα είναι διαθέσιμο. Περνάμε στο 7 που είναι η ομάδα εργασίας για τα παιδιά. Πρώτη συνεδρίαση στις 19 Οκτωβρίου διεξήχθη τότε. Δίνω στην Ελεονόρα τον λόγο για να μας πει ποια ήταν η έκβαση αυτής της εκδήλωσης. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπες η πρώτη μας ε, συνεδρία έλαβε χώρα στις 19 Οκτωβρίου και τα μέλη της ομάδας ε, αντάλλαξαν απόψεις ε, για το πώς θα, οργανωθεί, θα οργανωθούν οι εργασίες, να ζητήσουν το θέμα για την προφορική ερώτηση για το, το συμφέρον του παιδιού. Όπω επίση και την εφαρμογή της ενωσιακή νομοθεσίας για την προστασία των παιδιών ε, ε, από ε, τους υπαλλήλου Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέχρι τώρα η ομάδα εργασίας έχει αποφασίσει να ασχοληθεί με τα εξή θέματα. Πρώτον, την διεθνή απαγωγή παιδών, όπως επίσης υπηρεσία Jugendamt στη Γερμανία, η έγκριση χωρί την συγκατάθεση των γονιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ένα πάρα πολύ σημαντική συνάντηση που είχαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη συλλογή πληροφοριών, όπως επίσης τα κλεμμένα ε, νεογνά στην Ισπανία και, οποιαδήποτε θέμα μπορεί να προσθεθεί στην το χρόνο. Η ομάδα εργασίας θα συνέλθει πέντε φορές το 2016, Ιανουάριο, Απρίλιο, ε, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε έναν εξωτερικό εμπειρογνώμανα ανά συνεδρίαση. Το τέλος του 2016 θα κάνουμε έξεση σε έγγραφο εργασίε για τι ε, δραστηριότητε και τα πορίσματά μα. Όσον αφορά την προφορική ερώτηση για τα συμφέροντα των παιδιών σε διασυνοριακό επίπεδο στην Ένωση, τα, κράτη, τα μέλη τη ομάδα εργασία επεξεργάζονται το κείμενο και την τρίτη θα οριστικοποιήσουμε το κείμενο που θα πρέπει να συζητηθεί με τους συντονιστές της Γιούρη. Η τελική εκδοχή θα ε, εγκριθεί στην ε, συνεδρίαση του Δεκεμβρίου της Επιτροπής ΠΕΤΗ. Επίσης, ε, η Γενική Διεύθυνση Justice θα έρθει να συζητήσει το θέμα αυτό ε, και ανέφεραν ότι θα αναθεωρήσουν ε, το πρόγραμμα ε, της... Μας μίλησαν για το, την πρόθεσή τους να αναθεωρήσουν το νομικό πλαίσιο και τις σχετικές προτάσεις και ελπίζουμε οποιαδήποτε νέα στοιχεία προσθεθούν να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να αρχίσει η συζήτηση αν υπάρχουν συνάδελφοι που θα ήθελαν να σας θέσουν ερωτήματα για το θέμα αυτό ή αν έχουν γενικότερα σχόλια. Τατιάνα Ζδάνοκα και μετά ο Πίτερ Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που ε, υπάρχει αυτή η ομάδα εργασία. Θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε ε, επιτυχία στην προσπάθεια σας να προεδρεύσετε και να ε, καθοδηγήσετε τις εργασίες. δεν μπόρεσα να είμαι παρούσα στην προηγούμενη συνεδρίαση. Ήταν, η βοηθό, ήταν ο βοηθός μου παρόν και η πρότασή μου για ένα από τα θέματα έπρεπε να την υποβάλω στην Επιτροπή μας ε, όσον αφορά ε, τις ε, σκανδιναβικές χώρες Δανία, Σουηδία και Φινλανδία, την οποία υποστήριξε πολύ μεγάλη μη οργάνωση που, λαμβάνει, που δραστηριοποιείται στις σκανδιναβικές χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Νορβηγίας και αφορά τα παιδιά Ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε χώρο στην ημερήσια διάταξη στις συνεδριάσεις του επόμενου έτους. Θα προτιμούσα το συντομότερο δυνατόν, το Φεβρουάριο, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, αν μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε αυτήν, αυτές τις αναφορές που θα ήθελα να προτείνω και ελπίζω επίσης ότι θα εξεταστούν οι αναφορές αυτές και στην ομάδα εργασίας για τα παιδιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην ομάδα εργασίας, ε, επειδή είναι πολύ σημαντικό το έργο που αναλαμβάνει για το θέμα αυτό της Επιτροπής Αναφορών ε, για την εξέτασή του ε, για την ομάδα εργασίας. Είναι καλό ότι η ομάδα εργασίας καθόρισε σε ένα έτος να, έχει, να υποβάλει μια πρώτη έκθεση, να καταθέσει μια πρώτη έκθεση. Διότι τουλάχιστον βρισκόμαστε μπροστά σε δύο μεγάλα προβλήματα στην Επιτροπή Αναφορών. Πρώτον, σε αυτό το συγκινητικό από πλευράς ανθρωπιστικής θέμα να βρούμε Πού βρισκόμαστε και πού έχουμε αρμοδιότητες εμείς ως Ευρωπαίοι στο ευρωπαϊκό επίπεδο και πού δεν έχουμε αρμοδιότητες. Και όταν θα έχουμε καθορίσει την αρμοδιότητα στο ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο πιο κατεπήγον βρίσκεται στο να υπάρξουν κάποιες ε, τροποποιήσεις ή αλλαγές. Είναι σημαντικό το έργο αυτό που στο τέλος πρέπει να επιτελεστεί, νομοθετικό έργο δηλαδή από πράγμα του Ευρωκοινοβουλίου που πρέπει να προχωρήσει. Και δεύτερον, και ήταν και ένα βίωμα από την αποστολή μας διακρύβωση στο Λονδίνο να δούμε τι βρίσκεται ενδιάμεσα. Δηλαδή ευρωπαϊκή αρμοδιότητα των Βρυξελών και εθνική αρμοδιότητα από την άλλη πλευρά κρατών μελών. Αλλά όπως συμβαίνει με τους ανθρώπους υπάρχει ένα ενδιάμεσο πεδίο, ενδιάμεσο διάστημα. Πρέπει να βρούμε μια γλώσσα που αφενός να είμαστε συνεπείς, συνεπείς επί της ουσίας, αλλά παρόλα αυτά να μην περιφρονήσουμε και προσβάλλουμε την άλλη πλευρά. Για παράδειγμα, στην επαφή μας στην Βρετανία, παρότι είχαμε διαφορετικές απόψεις, υπήρχαν διαφορετικές απόψεις, να μπορέσουμε να δώσουμε συνέχεια. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην ομάδα εργασία, στο διαχωρισμό των ευθυνών και αρμοδιοτήτων και δεύτερον στο να βρεθεί ο τρόπο και η δυνατότητα σε σχέση με τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να υπάρξουν οι αναγκαίε αλλαγέ και προσαρμογέ που πρέπει να γίνουν. Ευχαριστώ. would you like to come? Κάποια σχόλια. να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την σωστή συνεργασία μαζί μας. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και νομίζω ότι ασχολούμαστε με το θέμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τη διαδικασία. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί προεδρεύεις αυτήν την ομάδα. Είναι βασικό το ότι δημιουργήσαμε αυτή την ομάδα εργασίας και ελπίζουμε να προχωρήσετε σύντομα στην, στα συμπεράσματά σας, στην κατάληξη μας περίπτωση της διαδικασίας. Γιατί έχουμε πάρα πολλές αναφορές. Ας περάσουμε στο 8 τώρα. Πρόκειται για την 0884-2014 της Σάρα Λαφουέντε Ερνάντες με πέντε υπογραφές για την παραβίαση από πλευράς της βελγικής κυβέρνησης του δικαιώματος παραμονής αλλοδαπού στο έδαφος του κράτους μέλους. Οι αναφερόμενοι είναι εδώ, θα τις δώσω αμέσως το λόγο. Όχι πάνω από πέντε λεπτά. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Πρώτα απ' όλα εξ ονόματος των συλλόγων και ενώσεων και εδώ στις Βρυξέλλες θα ήθελα να ευχαριστήσω την δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή και την ομάδα Ευρωβουλευτών που έδωσαν τη δυνατότητα να δοθεί συνέχεια σε αυτή την αναφορά τη δεχθήκατε και μας προσκαλέσατε να την παρουσιάσουμε εδώ σήμερα. Πιστεύω ότι όλοι εδώ γνωρίζουν τους όρους ε, ε στους οποίους ε, τοποθετείται αυτή η έκθεση ή η αναφορα σε σχέση με τις ε, απελάσεις και ότι 2.000, πάνω από 2.000 κοινοτικούς υπηκούς είχε απελάσει το Βέλγιο σε τέτοιου είδους απελάσεις που είχαν γίνει και το 2014 επίσης. Και μια και δεν υπάρχει αρκετός χρόνος θα παρουσιάσω τα ουσιοδέστερα σημεία που είναι τα πιο προβληματικά σε αυτή την βελγική πρακτική και την οδηγία 2004 κάθετος 38 για την ελεύθερη κυκλοφορία των κοινοτικών υπηκών και τα δικαιώματά τους που μου φαίνεται, μας φαίνεται ότι είναι πολύ προβληματική έτσι όπως έχει διατυπωθεί και λειτουργεί. Ε, καθορίζει όρους και ε, περιορισμούς για τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας. Ωστόσο πάνε πιο πέρα ακόμα οι διατάξεις του Βελγίου από ότι αυτά τα όρια που καθορίζει αυτή η οδηγία. Θέλαμε να τονίσουμε ότι στο Βέλγιο υπάρχει ένα σύστημα προσωπικών δεδομένων και διασταύρωσής τους μεταξύ των τοπικών αρχών που είναι εκείνε που είναι αρμόδιες για ε, κοινωνικά θέματα και και αυτή η διασταύρωση στοιχείων οδηγεί σε συστηματικούς ελέγχους για τους κοινοτικούς υπηκόους που επιθυμούν να έχουν την έδρα τους, να εγκατασταθούν στο Βέλγιο. Και η οδηγία ουσιαστικά ε, απαγορεύει τέτοιου είδους άμεσες εντολές απέλασης και γνωρίζει και αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή της αυτό το γεγονός. Αυτή η πρακτική επιπλέον παραβιάζει την ισότητα αντιμετώπισης των κοινοτικών υπηκόων στο Βέλγιο, διότι υποβάλλονται σε ειδικού ελέγχους από τη στιγμή που καταχωρούνται ως ε, εγκατεστημένοι στο Βέλγιο και υπάρχουν ε, ε, τέτοιου είδους έλεγχοι που δεν εφαρμόζονται στους ε, Βέλγους υπηκόους. Δεν υπάρχει λοιπόν ισότητα αντιμετώπισης και ταυτόχρονα έχουμε και παραβίαση των, της προστασίας προσωπικών δεδομένων διότι προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται από τις αρχές, τοπικές αρχές ώστε να, ε, ε, όταν υπάρχει αίτηση κοινωνικών επιδομάτων ακριβώς λοιπόν ε, χωρίς να υπάρχει έγκριση των ίδιων των ενδιαφερόμενων συντάσσονται οι εντολές απέλασης. Και έχουμε λοιπόν εδώ προβλήματα τα οποία τίθενται, διότι και οι αποφάσεις απέλασης καθώς επίσης και η διαγραφή ή να μην εγγράφονται σε τέτοια μητρώα, αυτό σημαίνει να υπάρχει έγκριση προηγούμενα των ενδιαφερομένων και όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει αναπερίπτωση να εξετάζονται σε σχέση με την κατάσταση αυτή στην οποία βρίσκονται αυτοί οι υπήκοοι και παραβιάζονται, οι αρχές της χάρτας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μας ανησυχούν λοιπόν οι πρόσθετες αυτές αρχές όροι και προϋποθέσεις και περιορισμοί από το Βέλγιο που δεν καθορίζονται με αντικειμενικά στοιχεία από πλευρά των βελγικών αρχών και έτσι υπάρχει αναπερίπτωση λοιπόν απόφαση και ε, εκτέλεση και δημιουργούνται πολύ μεγάλες ε, διαφορές μεταξύ των μεν και των δε διακριτικής ευχέρειας ε, στην εκτέλεση και εφαρμογή όλων αυτών. Και λέμε ότι αυτού του είδους οι αποφάσεις απέλασης ή άρνησης εγγραφής στο, στα Μητρώα Κοινοτικών Υπηκών είναι η κατάχρηση διακριτικής ευχέρειας και στην γραπτή απάντηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι ε, δεν δίνει απόλυτο, ε, δεν δικαιώνει απόλυτα αυτά τα επιχειρήματα. Και σε σχέση με το ότι κάποιος διαγράφεται από το σύστημα, αυτό έχει επιπτώσει στην καθημερινή του ζωή και δυσχεραίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ζωή του και την κατάστασή του στο Βέλγιο. Από την άλλη πλευρά θεωρούμε ότι η ίδια η οδηγία παραβιάζει έναν πυλώνα του κοινοτικού δικαίου όπως είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων υπηκών, της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας και απαγορεύεται η διακριτική αντιμετώπιση, ε, η επιβολή διακρίσεων διότι εδώ υπάρχει αποκλεισμός από την ελευθερία κυκλοφορίας μέσω ολόκληρης κατηγορίας κοινοτικών υπηκών, απλά και μόνο λόγω της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασής τους και πρέπει αυτό να αλλάξει οπωσδήποτε. Ε, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με την οδηγία και τα κράτη-μέλη, βλέπουμε σε ποια κατάσταση οδηγούμαστε, σε μια παρέκκληση, σε μια παρέκκληση, σε μια κατάσταση περιοριστική με ξενοφοβικές καταστάσεις και δράσεις σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά θα πρέπει να ανησυχήσουν και να κινητοποιήσουν τα ε, θεσμικά όργανα να δράσουν. Είναι υπεύθυνα τα θεσμικά όργανα για να μπορεί να διασφαλίζεται το δικαίωμα στην ελευθερία της κυκλοφορίας. Διακοινωτικά επί σειρά ετών, επί δεκαετίες και τώρα σε μια ε, φάση, σε μια συγκυρία οικονομικής ε, κρίσης ε, που θα έπρεπε να καταδειχθεί ότι πιστεύουν στην οικοδόμηση της Ευρώπης, κοινωνικής και ισότιμης Ευρώπης, παραβιάζουν αυτές τις αρχές. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Διαφορετικά δεν μπορεί να προχωρήσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα Υπάρχουν κατηγορίες και υποκατηγορίες λοιπόν κοινοτικών υπηκόων και υπάρχει και η παράνομη οικονομία στην οποία εξωθούνται η μαύρη οικονομία. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σε ευχαριστώ πολύ. Το πρόβλημα είναι ότι ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχει έρθει. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος του συγκεκριμένου υπαλλήλου ο κύριος πρόδρομος Μαυρίδης ή κάποιος άλλος. Έχετε το λόγο. And now, Μόλις έφτασε και η άλλη υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να αποφασίσετε ποιος θα πάρει το λόγο και ποιος θα εκφράσει την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα. I feel ε, συγγνώμη, δεν θέλουμε να σας πιέζουμε. Γι' αυτό mm. λοιπόν όλοι όσοι είσαστε στην αίθουσα ασχοληθείτε με τρυφερότητα με τον διπλανό σας. Κοιτάξτε, θα μιλήσω γαλλικά, η αναφορά είχε κατατεθεί στα γαλλικά. αμφισβητείται η απόφαση της Βελγικής Αρχής που αρνείται το δικαίωμα παραμονής σε Ευρωπαίους πολίτες. Ήδη από το 2014 τα μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν στο ότι η υπηρεσία αλλοδαπών είχε... Για, για μια στιγμή παρακαλώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από τους τεχνικούς να μας πει γιατί δεν γίνεται μετάφραση στα ισπανικά. Ζητώ συγγνώμη. Έχει σημασία βέβαια να ακούνε οι βουλευτές το τι θέλετε να πείτε. Λοιπόν, ξαναρχίστε. Επαναλαμβάνω, αμφισβητεί η αναφορά της αποφάσεις των βελγικών αρχών που αρνούνται το δικαίωμα παραμονή σε πολλούς Ευρωπαίους πολίτες. Ήδη από τον Ιανουάριο του 2014 πολλά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι η υπηρεσία αλλοδαπών του Βελγίου είχε εκδώσει 2.512 εντάλματα, ε, μάλλον απομάκρυνσης από το βελγικό έδαφος Ευρωπαίων πολιτών. Ξεκίνησαν κάποιες συζητήσεις με τις βελγικές αρχές γύρω από την υπόθεση αυτή σε σχέση με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αναφερόμαστε στο άρθρο 21 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίδει εγγυήσει σε όλα τα μέλη, σε όλους τους πολίτες το δικαίωμα να κυκλοφορούν και να εγκαθίσταται και να παραμένουν μάλλον. Το ίδιο άρθρο αυτό όμως λέει ότι ασκείται επί τη βάση των προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις συνθήκες και τις εφαρμοστικές αποφάσεις. Ήδη η συνθήκη ίδια δηλαδή προβλέπει ορισμένους περιορισμούς. Η οδηγία 2004-38 προβλέπει τις περιορισμούς αυτούς για τους πολίτες και τα μέλη των οικογένειών τους. Θέτει κάποιους όρους για παραμονή άνω των τριών μηνών. Για παραμονή άνω των τριών μηνών ε, τίθενται κάποιες προϋποθέσεις. Μέχρι τους τρεις μήνες υπάρχουν, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Μετά από τους τρεις μήνες έχουν δικαίωμα παραμονής εφόσον εργάζονται ή εφόσον αναζητούν θέση απασχόλησης ή έχουν επαρκή ε, έσοδα και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Η οδηγία διευκρινίζει επίσης ότι οι πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογένειών τους έχουν δικαίωμα παραμονής εφόσον δεν καθίστανται παράλογο βάρος ε, για το σύστημα το κοινωνικό της χώρας υποδοχής. Εφόσον οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν πληρούν λοιπόν τις προϋποθέσεις της οδηγίας, τα κράτη-μέλη μπορούν, μπορούν, δεν είναι υποχρεωμένα, να διαπιστώσουν ότι υπάρχει απουσία δικαιώματος παραμονής πλέον και ε, να αποσύρουν την δυνατότητα χορήγησης ε, κάρτας παραμονής και έτσι ε, δίδει, ε, εκδίδει αποφάσεις απομάκρυνσης από το βελγικό έδαφος και η βελγική διοίκηση. Αυτές οι αποφάσεις ε, γίνονται στα πλαίσια των εγγυήσεων τις οποίες καθορίζει η ίδια η οδηγία. Να εξηγήσω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από την άνοιξη του 2014 έχει ξεκινήσει έχει έρθει όπως είπα σε επαφή με τις βελγικές αρχές και συζητά την κατάσταση. Γιατί ακόμα και αν το Ευρωπαϊκό Δίκαιο επιτρέπει εκ των προτέρων σε ένα κράτος μέλος να διαπιστώσει το τέλος του δικαιώματος παραμονής ενός κοινοτικού αλλοδαπού, το σύστημα όπως λειτουργεί στο Βέλγιο παρουσιάζει ορισμένες φαιές περιοχές. Έχει ένα σύστημα αυτόματης ανταλλαγής δεδομένων ανάμεσα ε, στις υπεύθυνε ε, κοινωνικές υπηρεσίες, το ΙΚΑ ας πούμε το βελγικό, το ΣΕΠΑΕΣ και την υπηρεσία αλλοδαπών. Υπάρχει ένα αυτόματο σύστημα αλληλοενημέρωσης. Αν λοιπόν ένας ε, Ευρωπαίος πολίτης έχει τύχη κοινωνικών παροχών, τότε το όνομά του αποστέλλεται στην υπηρεσία αλλοδαπών, το οποίο μπορεί να ελέγξει αν ο συγκεκριμένος πολίτης εκπληρεί τις προϋποθέσεις παραμονής στην χώρα. Η συζήτηση λοιπόν με τις βελγικές αρχές συνεχίζεται, θέσαμε κάποιες ε, ε, ερωτήσεις και τέθηκε το θέμα κάποιων λεπτομεριών. Κάποιες συμβάσεις εργασίας, σαν παράδειγμα, δεν αναγνωρίζονται από τις βελγικές αρχές σαν γνήσιες και οι Ευρωπαίοι πολίτες που είχαν υπογράψει αυτές τις συμβάσεις έλαβαν εντολή απομάκρυνσης από το βελγικό έδαφος. Ενώ ε, υπάρχει η άποψη η οποία λέγει σύμφωνα με τις συνθήκες ότι είχαν ένα, τυπικά, ε, ένα τυπικό καθεστώς αναγνωρισμένο το οποίο θα τους επέτρεπε να παραμείνουν. Πάντως συνεχίζονται οι επαφές με τις βελγικές αρχές για τρία θέματα. Καταρχάς έλεγχος των διαδικασιών για την δημοσιοποίηση και γνωστοποίηση ε, της ε, λήξης του δικαιώματος παραμονής και επίσης για το θέμα της απομάκρυνσης από το Βέλγιο ε, ανέργων οι οποίοι είχαν εργαστεί στο Βέλγιο πριν πάρουν την ε, διαταγή απομάκρυνσης. Τίθεται λοιπόν το θέμα της ενημέρωσης της σωστής των Ευρωπαίων πολιτών και την δυνατότητα των Ευρωπαίων πολιτών να ε, ανταπαντήσουν στα επιχειρήματα των βελγικών αρχών τα οποία αιτιολογούν την απόσυρση του δικαιώματος παραμονής. Έχει ενδιαφέρον να πούμε εδώ ότι πρόσφατα ε, υπήρξε και μια προκαταρτική κατατέθηκε ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με το άρθρο 41 της Ευρωπαϊκής Χάρτας και αν εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη. Είναι θεμελιώδες το συγκεκριμένο ερώτημα γιατί το άρθρο 41 της Χάρτας ε, λέγει ότι υπάρχει δικαίωμα σε μια σωστή και εύρυθμη διοίκηση και αυτό ε, περιλαμβάνει το δικαίωμα κάθε προσώπου, κάθε πολίτη να μπορεί να εκφράσει την γνώμη του ε, προς τις αρμόδιες αρχές εάν ληφθούν εις βάρος του αρνητικές αποφάσεις. Και αυτό το δικαίωμα λοιπόν περιλαμβάνει και το δικαίωμα της πρόσβασης κάθε πολίτη στον φάκελο που τον αφορά, mm-hmm. στα πλαίσια βέβαια του σεβασμού της εμπιστευτικότητας κτλ και περιλαμβάνει επίσης την υποχρέωση για την συγκεκριμένη εθνική διοίκηση να τεκμηριώσει την απόφασή της. Η ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, νομίζω ότι θα καθορίσει τη συνέχεια των επαφών με τις βελγικές αρχές και εμείς εξαρτώμεθα από την ερμηνεία την οποία θα δώσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Νομίζω ότι λίγο πριν το καλοκαίρι θα μας δοθεί η, η απάντηση του δικαστηρίου και νομίζω ότι θα τακτοποιηθεί το θέμα πριν από το τέλος του 17 για να προστατευτεί από αμφιβολίες το δικαίωμα παραμονής. Πάντως εμείς συνεχίζουμε τις επαφές μας με τις βελγικές αρχές έτσι ώστε να εφαρμοστεί πλήρως η συγκεκριμένη οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα και διεξοδικότατη ε, απεικόνηση της κατάστασης παρά το γεγονός ότι ήσασταν ε, λίγο αμήχανοι όταν μπήκατε στην αίθουσα. Η κυρία Βαλίνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς υποστηρίζουμε απόλυτα αυτή την αναφορά. Θεωρούμε ότι υπάρχει παραβίαση της οδηγίας από πλευράς βελγικής νομοθεσίας. Και λέμε γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει αυτή η παραβίαση. Πρώτον, επειδή υπάρχει συστηματικός έλεγχος των όρων εγκατάστασης και επειδή υπάρχει απουσία ισότητας αντιμετώπισης σε σχέση με τους υπηκόους κρατών μελών και θεσπίζονται μέτρα αυτόματα απέλασης αλλοδαπών όταν χάνουν την απασχόλησή τους, την υποτροφία τους ή κάτι σχετικά παρόμοιο. Και επιπλέον εδώ υπάρχει η αρνητική μεταχείριση σε σχέση με τους όρους οικονομικούς που απαιτούνται και που καθορίζονται με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τα μέλη μιας οικογένειας αλλοδαπών, σε σχέση με άλλους υπηκόους. Παραβιάζονται πολλά άρθρα της ε, Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, ένα και μόνο παράδειγμα, το 15.2, η ελευθερία αναζήτησης απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη-μέλη της, μέλη της. Στα κράτη του Νότου έχουμε υψηλότατα ποσοστά ανεργίας, την κρίση, την ε, περίοδο λιτότητας που υποχρεώνουν τους νέους μας να αναζητήσουν απασχόληση αλλού. Υπενθυμίζω το 50% της ανεργίας των νέων στην Ισπανία. Είναι υποχρεωμένοι οι ναι, να αναζητήσουν μέλλον αλλού που δεν βρίσκουν στο, το μέλλον αυτό στη χώρα τους. Περνάνε λοιπόν σε άλλη χώρα και έχουμε εδώ όταν ε, δεν γίνονται δεκτοί και απελάβνονται παραβίαση αυτής της αρχής ελεύθερης κυκλοφορίας. Εδώ οι πολίτες κρίνονται από τα πόσα μηδενικά έχει ο λογαριασμός τους στην τράπεζα, πόσα χιλιάρικα έχουν ε, στην, ε, στο λογαριασμό τους. Παραβίαση λοιπόν όλων των αρχών και του άρθρου 9 της μη αρνητικής ε, μεταχείρισης των μη διακρίσεων όσον αφορά την υπηκότητα. Υπάρχει έρευνα σε σχέση με τις βελγικές αρχές όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ολοκληρωθεί αυτός ο έλεγχος ακόμα. <clears throat> Δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε στα τέλη του 17 για να δούμε τι γίνεται με αυτά τα άτομα που απελάβνονται. Λοιπόν, επί ένα χρόνο θα βρίσκονται, θα εκκρεμούν οι υποθέσεις και τι θα γίνεται, που θα, σε ποια κατάσταση θα βρίσκονται. Γι' αυτό θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σοβαρό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τηρεί τις βασικές και θεμελιώδεις αρχές για τις οποίες δημιουργήθηκε και στα θεμέλια των οποίων δημιουργήθηκε. Και η κρίση οδηγεί στο να υπάρχει ρατσισμός, διακριτική μεταχείριση σε μια Ευρώπη που δεν θέλουμε να έχει αυτό το πρόσωπο και δεν την αναγνωρίζουμε με αυτά τα χαρακτηριστικά. Το πρόβλημα, το θέμα είναι τόσο σοβαρό και τόσο βαθύ που εμείς θα ζητούσαμε προφορική ερώτηση στην Ολομέλεια να κατατεθεί με ψήφισμα δεν είναι δυνατόν να έχουμε τον χρόνο λοιπόν να ακούσουμε όλες τις επεξηγήσεις εδώ. Θέλουμε μια προφορική ερώτηση και να απαντηθεί αυτή η ερώτηση από την Επιτροπή και να γίνει αυτή η συζήτηση και να μας πούν τι σκέπτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά τα μέτρα και πώς σκέπτεται να επιλύσει το πρόβλημα αυτών των ατόμων. Δεν μπορούμε να δεθούμε τέτοιες αρνητικές μεταχειρήσεις λόγω οικονομικών όρων και προϋποθέσεων όχι μόνο σε σχέση με ε, τα, την αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων αλλά και των εμπορευμάτων που αντιμετωπίζονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλει κανένας άλλος να πάρει το λόγο. Μήπως ε, θέλει κανείς άλλος συνάδελφος να πάρει το λόγο. Οπότε ξαναδίνω το λόγο στην ε, Σάρα Λαφουέντερνάντες. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Muchas Σας ευχαριστώ πολύ. Κρίμα είναι που η εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής δεν παρίσταται όταν ε, κάναμε την παρέμβασή μα. Εκφράζουμε βαθύτατη θλίψη γι' αυτό. Αλλά επίση και ότι, γιατί δεν υπήρξαν σχόλια από άλλου ευρωβουλευτέ γι' αυτό. Ένα θέμα τόσο ευαίσθητο και σοβαρό και που έχει τόσο άμεσες επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, για τους πολίτες, ιδιαίτερα για τους πολίτες των κρατών του Νότου της Ευρώπης, αλλά και για τον, τους τη της Ανατολικής Ευρώπης, κρατών της Ανατολικής Ευρώπης, που με τον ίδιο τρόπο πλήττονται. Θα έπρεπε να γίνει μεγαλύτερη συζήτηση και μας εκπλήσει το δεν έγινε αυτό σε σχέση με την Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την απάντηση που δόθηκε από πλευράς Ευρωβουλευτού που πραγματικά θα ήταν ενδιαφέρον η κοινοβουλευτική σας επιτροπή να συνέχιζε τη συζήτηση αυτού του θέματος και να μπορούσε με προφορική ερώτηση να καταλήξει στην Ολομέλεια. Δεν ξέρω με ποια διοικητική διαδικασία για την Ολομέλεια να, για να μπορέσει να, να λάβει υπόψη σοβαρά το θέμα αυτό ώστε το Κοινοβούλιο να αναλάβει επιτέλους κάποια πρωτοβουλία και να τοποθετηθεί με σαφήνεια υπέρ μιας ε, κοινωνικής Ευρώπης και των δικαιωμάτων των πολιτών ε, που πλήττονται εδώ άμεσα και εξίσου πιστεύω ότι και συμμερίζομαι την ανησυχία της Ευρωβουλευτού που παρενέβη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι υπάρχει μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που εκρεμεί για το θέμα του αν εφαρμόζεται ή όχι η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για τους υπηκόους αυτών των κρατών. Αναμένουμε, αν και περιμένουμε και συζητάμε εδώ και ένα χρόνο, αλλά θα έπρεπε άμεσα να ληφθεί απόφαση γιατί πλήττονται εδώ πάμπολοι Ευρωπαίοι, πάρα πολλοί άνθρωποι και το ευρωπαϊκό εγχείρημα πλήττεται επίσης. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να σας πω ότι η εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, προτίθεται να σας μιλήσει αμέσως ε, μετά το τέλος του θέματος αυτού του σημείου της μηνύσης διάταξης. Νομίζω ότι αυτή η επαφή μαζί της θα είναι νομίζω πολύ σημαντική και χρήσιμη για σας. Κύριε Μαρτά, έχετε το λόγο. Εγώ απλώς ε, θα ήθελα να σχολιάσω με απασχολεί πολύ αυτό το θέμα. Δεν θέλω να παίρνω το λόγο σε συζητήσει οι οποίε έχω καθυστερήσει. Λυπάμαι κιόλα, αλλά είναι πολύ ευαίσθητο αυτό το θέμα και επειδή δεν γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες της ε, αιτιολόγησης, όταν όμως διαβάζω την αναφορά, ε, ανεξαρτήτως λόγου είναι αδύνατον ένα, μέλος της, ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύει τη διαμονή ενός Ευρωπαίου υπηκόου στο έδαφος του. Πρέπει οπωσδήποτε να αποτελέσει πραγματικότητα η ελευθερία ε, κυκλοφορίας των πολιτών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην είναι απλώς μια θεωρία Ευχαριστώ. Ξαφνικά όλοι θέλουν το λόγο. Κυρία Εύη και μετά νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι φυσικά και συμφωνώ με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης αναφοράς. Είναι απίστευτο, όπως είπε και ο συνάδελφος Μαρτά, η Ευρώπη να βασίζεται στην ιδέα της ελεύθερης διακίνησης, κυρίως των εμπορευμάτων. Και, όχι, και δεν σέβεται στην ουσία τα δικαιώματα των πολιτών και δημιουργεί εμπόδια στα πρόσωπα, στους πολίτες και στα δικαιώματά τους. Νομίζω ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε με την οδηγία αυτή, πρέπει να μείνει ανοιχτή και να στηρίξουμε όσο μπορούμε περισσότερο τους αναφερομένους. Ευχαριστώ ε, πολύ. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, οπότε μπορώ να συμπεράνω ότι βεβαίω θα παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Θα αποστείλουμε επιστολή στις βελγικές αρχές ε, ζητώντας ε, ακριβέστερες πληροφορίες και επίση δεδομένων όσων υπόθηκαν από τους συναδέλφους ε, βάσει του άρθρου 9 ε, και του άρθρου 21 της Συνθήκης για τη Λειτουργία ε, της Ένωσης που εξασφαλίζει την ελευθερία μετακίνησης και διαμονής σε άλλο κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα να ρωτήσω τις βελγικές αρχές ποιες είναι ακριβώς αυτές οι ε, διαδικαστικές εγγυήσεις, ε, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα του εισακούεσθε ε, και ποια είναι η επιχειρηματολογία τους, εν πάση περιπτώσει, για το θέμα αυτό πριν απελάσουν κάποιον, πριν τον απομακρύνουν από την επικράτειά τους. Τώρα, η πρόταση της κυρίας Βαλίνα για προφορική ερώτηση και ψήφισμα, όπως όλοι γνωρίζουμε αυτό πρέπει να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη συνεδρίαση των συντονιστών και να το ξανασυζητήσουμε και να δούμε πώς θα, αποφασί... πώς θα προχωρήσουμε. Το σημειώνουμε, θα το σημειώσει και η γραμματεία και θα δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε τον καλύτερο δυνατό ε, τρόπο ακολουθώντας τις διαδικασίες. Είναι γεγονός πάντως ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης για τους πολίτες της Ένωσης που είναι μια βασική αρχή της που δεν πρέπει να παραβιάζεται ποτέ. Αυτό είναι, αυτή είναι η ουσία αυτής της Επιτροπής και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε πολύ ομόφωνοι ως προς αυτό. Να σας επιστήσω και την προσοχή στο ότι αυτή η Επιτροπή, η ΠΕΤΗ, από κοινού με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, δρομολόγησαν μία μελέτη για την ελεύθερη κυκλοφορία ε, από το ε, τμήμα μελέτης η οποία θα μας ε, παρασχεθεί το 2016 Πραγματικά είναι πολύ επίκαιρο αυτό να δούμε πώς συνδέονται διάφορα πράγματα μεταξύ τους, πώς ε, ακριβώς συνδέονται ώστε να δημιουργούν αυτήν την εικόνα και να έχουμε και μια λεπτομερή εικόνα της κατάστασης. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την αναφέρουσα, την κυρία Κερνάντες και να σας εκφράσω την πλήρη υποστήριξή, μας, της Επιτροπής μας ε, για ε, την αναφορά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν τόσο ακριβείς και τόσο ε, σαφής στην ε, περιγραφή των ε, ε, δεδομένων. Σας καλώ να έρθετε σε διάλογο με την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό κατά τις ερχόμενες ημέρες. Ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. You know, today is a... Είναι η τυχερή μας μέρα. Έχουμε χρόνο. Μας μένει χρόνο. Δεν συμβαίνει ποτέ αυτό. Λοιπόν, 10 λεπτά διάλειμμα άρα. Ελπίζω να επιστρέψουμε όλοι στις 11.30 ακριβώς. 11.30 να καθόμαστε, ώστε να μπορούμε να έχουμε ε, την κοινή συνεδρίαση με τη ΛΥΜΠΕ για την ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για ε, την έρευνα ε, ιδία πρωτοβουλία για, τη front, για το Frontex. Ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ επιστρέψτε σε 11.30. Okay, back. I hope Λοιπόν, ε, Ελπίζω η διακοπή σύντομη να ήταν ευχάριστη και καρποφόρα. Και να καλωσορίσω την Κίνγκα Γκάλ που μόλις τώρα κάθεται και όλους τους συναδέλφους από τη Λίμπε. Είναι σημαντικό που έχουμε αυτή την κοινή συνάντηση. Σας καλωσορίζω λοιπόν σήμερα στη δεύτερη κοινή συνάντηση για την έκθεση των Ombudsman ε, για το, του Ομπουτσμαν μάλλον συγγνώμη, για το Frontex. Έχουμε λάβει 199 τροπολογίες. Αμέσως μετά από αυτή τη συνάντηση οι Σκιώδης σε συνεργασία με τους Σκιώδης θα έχουν μια συνάντηση για την έβρεση πιθανών συμβιβαστικών προτάσεων τροπολογιών. Η τροπολογίες αυτές ε, θα πρέπει να κατατεθούν εγκαίρως στην αγγλική γλώσσα. Έχουν μεταφραστεί όμως ήδη από χθε ε, και στις άλλες γλώσσες, όσες κατετέθηκαν μάλλον σε άλλες γλώσσες, μεταφράστηκαν και ε, έχουν διανεμηθεί στο έγγραφο χτες το απόγευμα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο εδώ στη συμπροεδρό μου, την Κίνγκα Γκάλα από τη Λίμπε, και μετά στους εισηγητές και μετά στους σκιώδεις εισηγητές και αργότερα στα υπόλοιπα μέλη. Κίνγκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θεσίλια. Μία σύντομη παρατήρηση. Είχαμε μια πολύ θετική πρώτη συζήτηση στην χθεσινή προκαταρκτική συνάντηση Υπήρξε σωστή συνεργασία ανάμεσα στους δύο εισηγητές, θα συνεχιστεί η συνεργασία αυτή όταν συζητηθούν αργότερα σήμερα και οι δυνατότητες τροπολόγησης. Ας περάσουμε λοιπόν στους εισηγητές χωρίς άλλη καθυστέρηση, εισηγητές, Σκιώδης και τα υπόλοιπα μέλη. Ευχαριστώ. Εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών είναι μεγάλη τιμή να συνεργάζομαι με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ γιατί εμείς δεν είμαστε νομοθετική επιτροπή, η Επιτροπή Αναφορών δεν είναι νομοθετική επιτροπή και πρέπει να στραφούμε προς τις νομοθετικές επιτροπές για να μπορέσουμε με επικοδομητικό τρόπο ε, να δουλέψουμε. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μέτσολα, πρώτη εισηγήτρια. Ευχαριστώ Σεσίλια, ευχαριστώ Κίνγκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ για το μεγάλο ενδιαφέρον που καταδείχθηκε από πλευρά σας και μπορώ να σας διασφαλίσω ότι από κοινού με ε, τον συνάδελφό μας είχαμε εξαιρετική συνεργασία για αυτή την έκθεση. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να συμπεριληφθούν όλοι από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στους συμβιβασμούς που συμφωνήσαμε. Και χθε μας εξέπληξε θετικά, με ιδιαίτερα θετικό τρόπο, το υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε και εκφράστηκε για αυτή την έκθεση. Και μπορώ να σας πω ότι περίπου 200 τροπολογίες κατατέθηκαν από ευρωβουλευτές από το σύνολο του πολιτικού φάσματος των ε, πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου. Και ακριβώς επειδή είχαμε ζητήσει και εσείς είχατε καταδείξει την υπομονή και δεχθήκατε το ότι δηλαδή θα έπρεπε να είναι οι τροπολογίες στα αγγλικά, μπορούμε λοιπόν να έχουμε τις τροπολογίες αυτές και να γνωρίζουμε το τι συμβαίνει με αυτές τις τροπολογίες συγκεκριμένα. Εισαγωγικά αυτά πήραμε τροπολογίες που συμπεριλαμβάνουν περαιτέρω θετικές αναφορές όσον αφορά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό ότι η υπηρεσία έλαβε υπόψη ε, η Frontex ε, τις συστάσεις που εκφράστηκαν από τον Ευρωπαίο Διασμεσολαβητή. Επίσης ε, και για την διαφάνεια όσον αφορά μηχανισμούς εξέτασης παραπώνων και τα θέματα που αφορούν την, ε, το, την Frontex άμεσα για ε, υποθέσεις που αφορούν τα κράτη-μέλη και ε, διευκρίνησε ότι η Frontex θα χρησιμοποιήσει τις αναγκαίες εκείνες, τα αναγκαία ειχέγγυα που θα ισχύουν και θα λειτουργούν όταν θα υπάρχουν προσωπικά παράπονα, παράπονα ατομικά τα οποία θα εκφράζονται ώστε να μπορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα, η υπηρεσία, ο οργανισμός θεμελιωδών δικαιωμάτων να μπορέσει να λειτουργήσει και να δράσει εξετάζοντας τα παράπονα και τις προσφυγές που θα έχουν ασκηθεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διαφορετικά δεν θα μπορέσει η Frontex να υλοποιήσει αυτές τις συστάσεις μέσω αυτού του μηχανισμού. Και τέλος, ε, λάβαμε διάφορες ε, τροπολογίες από διάφορες, ε, διαφορετικές ομάδες και ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε στην προστασία ιδιαίτερων ομάδων όπως των ασυνόδευτων ανηλίκων παιδιών. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσω το λόγο τώρα και στη Σκά Κέλλερ που είναι στην εισηγήτρια. Με πολλή αγωνία περιμένουμε να σας ακούσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και, στην, ε, και τη Ρομπέρτα για την πολύ καλή συνεργασία. Χθε ήταν η προθεσμία, χθε στι 12 το μεσημέρι, για την υποβολή τροπολογιών. Ε, πάρα πολλοί κόσμο έμεινε ξύπνιο ω αργά για να βρεθούν συμβιβαστικέ λύσει. Θα γίνει μια συνάντηση των σκιωδών εισηγητών μετά την τωρινή συνεδρίαση. Θα ε, εξετάσουμε διεξοδικά όλε τι συμβιβαστικέ τροπολογίε που προτείνουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν για παράδειγμα τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες ε, που ε, κάποιες ε, ομάδες τόνισαν ιδιαίτερα. Νομίζω ότι είναι πολύ ε, παρόμοιες οι απόψεις μας, ε, ε, οι, ποιοι συμμετέχουν στις υπηρεσίες της Frontex και τι ακριβώς θα γίνει με τους συνοριοφύλακες, όπως και τις ανώνυμες προσφυγές που κάποιοι τους, τις απέρριψαν, κάποιοι τις πρότειναν. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Όσον αφορά τις τροπολογίες για τις γλώσσες που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για το φόρουμ αλλά και για τις πληροφορίες, ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα, του, θα μας βρει όλους σύμφωνος. Το θέμα επίσης της αναγνώρισης ε, των, ε, του της τακτοποίησης των, του προσωπικού. Άλλα, άλλοι συμβιβασμοί που θα μπορούσα να σας ε, τονίσω είναι το θέμα της συνεργασίας, για παράδειγμα, μεταξύ των δικαιωμάτων ε, ε, και ε, των δυνατών, των πιθανών προσφυγών τις οποίες μπορεί να προβεί η Frontex όταν υπάρχουν σοβαρές ε, παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, η επαρκή στελέχωση και η επαρκή χρηματοδότηση είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε και με τους υπόλοιπους και όδης εισηγητές. Το θέμα των ευάλωτων ομάδων νομίζω ότι μας βρίσκει όλους σύμφωνους, πώς μπορούμε δηλαδή να ε, παρεμποδίσουμε την παραβίαση δικαιωμάτων με βάση το φύλλο λάβαμε κάποιες τροπολογίες και σχετικά. Σε γενικές γραμμές έτσι έχουν τα πράγματα. Για αυτούς τους τομείς που ανέφερα ε, σε αδρές γραμμές αναζητούμε συμβιβασμούς. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς ε, γιατί έχουμε 200 τροπολογίες. Ε, η ψηφοφορία θα γίνει την Δευτέρα, οπότε μόνο μερικές μέρες έχουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας, για, για τη συνεργασία σας ε, κατά τις επόμενες ημέρες αλλά και για τις τροπολογίες σας. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ε, οι συνεισηγήτριες ε, θα εξετάσουν τις τροπολογίες αυτές. Τότε, τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο σε όσους και οι συζητητές θέλουν να πάρουν το λόγο. Με χαρά αναμένουμε τη συνεισφορά σας. Κύριε Μαρτάν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Βλέπουμε ότι είναι μια έκθεση η οποία είχε ως αποτέλεσμα πολλούς προβληματισμούς και πολλές τροπολογίες. Ε, θέλουμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία του Frontex. Συμφωνώ με την τροπολογία που αφορά την καλύτερη αναγνώριση και την ε, ε, εξέταση του προβλήματος των πιο ευάλωτων ομάδων, για παράδειγμα των εγγύων γυναιτών. Καταλαβαίνω ότι η Frontex έχει ε, πρόβλημα με την αποδοχή των ανώνυμων προσφυγών, οπότε επειδή είναι ένα θέμα που αποσχολεί πολλά κράτη-μέρη πρέπει να μπορέσουμε να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν. Θα ήθελα επίσης να ενθαρρύνω τη συνεργασία με ε, το την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης ε, για το Άσυλο. Αυτά ήθελα να πω σε γενικές γραμμές. Όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα θα έλεγα ότι είναι ένα κείμενο το οποίο είναι αρκετά ισορροπημένο και θα βελτιώσει το τα δικαιώματα των ε, μεταναστών και των προσφύγων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Νάγκη. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για το έργο που επιτελέστηκε και για την προετοιμασία ενός καλού εγγράφου. Και σας ευχαριστούμε και για τις 200 ε, τροπολογίες. Ε, πρέπει να τονιστεί ότι είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί ένας λειτουργικός μηχανισμός επίλυσης ε, παραπώνων για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες όταν υπάρχει κάποια παραβίαση. Για έναν λειτουργικό μηχανισμό θα χρειαστούμε, θα χρειαζόμαστε και αναγκαία κονδύλια, χρηματοδότηση δηλαδή και ενδυνάμωση της Frontex που είναι πολύ σημαντικές πτυχές. Επίσης, δεν πρέπει να δημιουργηθεί δυσλειτουργικό γραφειοκρατικό βάρος για αυτή την υπηρεσία που είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να λειτουργήσει μια και έχει τόσες πολλές αρμοδιότητες, ιδιαίτερα στην ε, λειτουργία αναχέτησης, στις δράσεις ε, pushback αναχέτησης ε, μέσω των παρεμβάσεων και με τα παράπονα που υπάρχουν πρέπει να υπάρξει ένας λειτουργικός μηχανισμός ε, αντιμετώπισης τους ε, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το έργο από πλευράς υπηρεσίας αλλά και ο μηχανισμός αυτός να είναι λειτουργικός. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ έχουμε αυτές τις τροπολογίες ε, στις, μπροστά μας ε, στο τραπέζι και είναι πολλές ε, εκτενείς και διεξοδικές. Καμιά φορά είναι ανησυχητικό ότι η κατάσταση στα κράτη-μέλη με διαφορετικό τρόπο αντιμετωπίζεται. Ακόμα και τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με διαφορετικό τρόπο κρίνονται και αξιολογούνται. Και γι' αυτό πρέπει να διαπιστώσουμε και να πούμε ότι κυρίως η κατάσταση για τα παιδιά και τις γυναίκες είναι πολύ ανησυχητική. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης και θα προσπαθήσω από πιο κοντά να τα εξετάσω και να τα συζητήσουμε και σε σχέση και με τους κοιόδης εισηγητές. Σε αυτό το ζήτημα χρειαζόμαστε σαφέστατες διατυπώσεις, ώστε τουλάχιστον τα παιδιά και οι γυναίκες να προστατεύονται επαρκώς. Κυρία Ξεκινώντας θέλω να ευχαριστήσω τους δύο συνεισηγητές αλλά και τους σκιώδεις ε, για την συνεισφορά τους. Υπήρξε πολύ ενδιαφέρον για την έκθεση αυτή. Οι προτάσεις ε, έτσι όπως έχουν κατατεθεί μπορούν να ε, βοηθήσουν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ευάλωτων κατηγοριών ε, και τον ρόλο των Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Υπηρεσιών. Δύο βασικές προτάσεις τις οποίες καταθέτω εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας. Καταρχάς οι τροπολογίες ε, ε, έχουμε, καταθέσει προς την κατεύθυνση αυτή. Ε, υπάρχει μια έκκληση γενικά ε, έτσι ώστε να υπάρξει ενημέρωση για τα παράπονα και τις διαμαρτυρίες σχετικά με το Frontex και θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι δεν πρόκειται για ένα θέμα ε, απλά του να προσπαθήσουμε να ονοματίσουμε και να κατηγορήσουμε αλλά να εντοπίσουμε τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να εργαστούμε σκληρότερα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στα παράπονα αυτά, στις διαμαρτυρίες αυτές και να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε σωστά το προσωπικό έτσι ώστε να βελτιώσει τη συμπεριφορά του. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους υπάρχοντες, τις υπάρχουσες μάλλον δυνατότητες για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Γι' αυτό λοιπόν έχουν κατατεθεί οι τροπολογίες ε, οι τροπολογίες από πλευράς μας ε, και σε σχέση με ό,τι αφορά στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα επιδιώξουμε τη βέλτιστη πρακτική ε, με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδιαίτερα σεβόμενοι τα δικαιώματα των ευάλωτων κατηγοριών όπως των ασυνοδεύτων ανηλίκων. Υπάρχει ανάγκη εμείς να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις στην παρούσα φάση των μεταναστευτικών ρευμάτων των τόσο ισχυρών και να ορίσουμε σωστά τις ευθύνες ε, ε, και επίσης τις αρμοδιότητες του Frontex. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους λοιπόν και όλους τους συναδέλφους για την υποστήριξή τους. Η Εύη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια ή τις εισηγήτριες μάλλον για την εξαιρετική τους δουλειά. tra tutti il fatto che Frontex essendo, essendo Μιλάμε για μια ευρωπαϊκή υπηρεσία και γι' αυτό είναι βασικό όλες, όλοι υπάλληλοι οι οποίοι εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και εργάζονται για αυτήν να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι μια βασική αρχή πάνω στην οποία θα έλεγα βασίζεται η ίδια η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να υπογραμμίσω εδώ την ανάγκη να υπάρξει ένας ανεξάρτητος ε, μηχανισμός και γι' αυτό προτείνουμε έναν μηχανισμό στον οποίο θα καταντήθενται οι καταγγελίες με ανεξάρτητο και προστατευόμενο τρόπο και όλα τα αιτήματα τα οποία θα παρουσιάζονται και όλες οι καταγγελίες οι οποίες θα γίνονται να θεωρούνται αποδεκτές εφόσον βέβαια εκπληρούνται κάποιες βασικές κάποια βασικά χαρακτηριστικά, κάποιες βασικές ιδιότητες. Ο μηχανισμός που θα ισχύσει θα πρέπει να καθιστά τη διαδικασία όσο περισσότερο ανεξάρτητη γίνεται. Τώρα, για τους υπαλλήλου, για τους εκπροσώπους, σε πάση περιπτώσει της Frontex ή για τους ε, ε, αποσπασμένους εθνικούς υπαλλήλου, εφόσον διαπιστωθεί μια σοβαρή παράληψη, παραβίαση από μέρους τους, θα πρέπει να απομακρύνονται αμέσως από το Frontex, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα βέβαια και έφεσης και η δυνατότητα οι καταγγελίες να κατατίθενται και από τρίτους στη συγκεκριμένη περίπτωση από μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Θα συμφωνήσουμε λοιπόν με τις τροπολογίες οι οποίες ε, θέλουν να υπάρξει μια καταλογοποίηση των καταγγελιών αυτών και θα μας επιτρέψει αυτό να έχουμε δεδομένα στατιστικά που θα βοηθήσει με τη σειρά του την αξιολόγηση των καταγγελιών αυτών. Ένα τελευταίο σημείο αφορά την δημοσιοποίηση της ύπαρξης αυτού του μηχανισμού είτε μέσω των εθνικών αρχών είτε μέσω των υπηρεσιών της ίδιας της Frontex. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Κούνεβα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ευρώπη και η ηγεσία τη είναι απλώ λόγο ένοχη από την τραγωδία που εξελίσσεται στο Αιγαίο και σε όλο το Μεσόγειο. Και ένα από του λόγου που είναι ένοχη είναι η ίδια η Frontex η Frontex, ο πρώτος πανευρωπαϊκός φράχτης, πριν και μίσον φράχτες σχεδόν όλα τα σύνορα της Ευρώπης. Η Frontex ήταν και παραμένει η δύναμη που σπρώχνει τους επελπισμένους πρόσφυγες στους επικίνδυνους δρόμους που τους ανοίγουν οι διακινητές. Ευθύνεται άμεσα ή έμεσα εκατοτάδεν των άσως πρόσφυγων. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτε πιο υποκροτικό από το να ορίσουμε την Frontex υπεύθυνη για την προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων που η ίδια πρώτη παραβιάζει. Το δικαίωμα των πρόσφυγων και των μετανάστη να καταγγέλει ό,τι γίνεται σε βάρος του μπορεί να ασκείται πραγματικά μόνο σε έναν ανεξάρτητο μηχανισμό καταγγελιών που θα λειτουργεί με την ευθύνη της Είπα της αρμοδιότητας το ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και άλλων ανεξάρτητων ανθρωπιστικών οργανώσεων. Είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στους χιλιάδες απελπισμένους. Είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των χιλιάδων νεκρών πρόσφυγων. Στο Λέσβο δεν υπάρχει πια χώρος να τάψουν τους πρόσφυγες. Είναι γεμάτο το νησί. Δεν υπάρχει χώρο ούτε να περπατήσουν οι άνθρωποι από τάφους μεταναστών και τα ψυγεία πια είναι γεμάτα. Αλλιώς είναι σαν να βάζουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα αν ορίσουμε το Frontex να ελέγχει την κατάσταση. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Δεν ήξερα ότι είσαστε Ελληνίδα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Um, now I would like to give the floor to η Αντζέλικα Μελινάρ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα μία ακόμη φορά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στις εισηγήτριες για την εργασία τους. Δυστυχώς δεν είχα χρόνο να εξετάσω όλες τις τροπολογίες, γιατί χθες μόλις τις ε, λάβαμε, χθες το βράδυ. Αλλά φυσικά θα γίνει μία ανάλυση όλων των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. Θα ήθελα να τονίσω όμως τα εξή ότι ο μηχανισμό θα πρέπει να είναι σαφή και για τι δύο πλευρέ και για του υπαλλήλου του Frontex αλλά και για τα πιθανά θύματα. Πρέπει να είναι σαφή ποιος θα χρησιμοποιεί το μηχανισμό και για ποιο λόγο οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο, οι ευάλωτες ομάδες όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και ε, οι έγκυες γυναίκες πολύ συχνά ε, είναι θύματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους αλλά ίσως αυτός ο μηχανισμός να μην είναι ο κατάλληλος για να ε, ληφθούν υπόψη όλες οι καταγγελίες γιατί το θύμα θα χάσει χρόνο εάν δεν καθοδηγηθεί στις σωστές αρμόδιες αρχές. Και επίσης θα ήθελα να αποφευθεί το ε, με ε, λιώδες δικαίωμα ε, θα ήθελα να αποφευχθεί η παραβίαση της θεμελιώδους δικαιώματος για καταγγελία η Ουγγαρία και οι κάτω χώρε μα υπενθυμίζουν συνεχώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα αποτελεσματικό μηχανισμό το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο, και εγώ ευχαριστώ. Θέλει κανεί άλλο να πάρει το λόγο. Να δώσω το λόγο και πάλι στις εισηγήτριες, πρώτα στη Σκακέλερα αυτή τη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω, γιατί πρέπει να βρούμε συμβιβαστικέ λύσεις τώρα, εξετάζοντας τροπολογίε και ελπίζω να τα καταφέρουμε στη συνάντηση των σκιωδών. Ρομπέρτα, μήπως θέλεις να προσθέσεις τίποτα? Απλώς να ευχαριστήσω όλους σας για τη ε, συνεργασία σας. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν ευρύτερη συνένεση για την έκθεση αυτή. Μάλιστα, καταπληκτικά. Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε από αυτού. Η επόμενη κοινή συνεδρίαση θα λάβει χώρα τη Δευτέρα στις 6. Μην ξεχάσετε να φέρετε τότε τις κάρτες σας για την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά για σήμερα. Τη Δευτέρα ξανά.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 dans une manière anonyme peuvent faire cela avec une organisation ONG, par exemple. Okay, I will later then explain that in English. That would be perfect if you can do that. That's what I was suggesting. Okay, here goes my French lesson. Merci, merci. Thank you.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 Okay.